Good morning, dear colleagues. I wish... Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Με πολλή επιτυχία, πολλές επιτυχίες. Σε αυτή χρονιά. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας και γι' αυτό σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω ότι λόγω των ε, προβλημάτων χώρου, έλλειψη δηλαδή θαλάμων, δεν έχουμε φινλανδική, εσθονική και ε, μαλτεζική διερμηνία για το πρωί και φινλανδική, εσθονική για το απόγευμα. Δεν είχαμε αρκετούς θαλάμους. Επίσης μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 6 ψηφοφορία για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφαλεία δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Έχει αναβληθεί η ψηφοφορία τη έκθεση του κ. Σλίτσερ για τι 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Στην προσοχή μα συνεδρίαση και αν δεν έχετε αντιρρήσει, ε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με τι τροποποιήσει τη. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών τη της συνεδριάσεως 8 και 9 Ιουλίου 2013, 5 Σεπτεμβρίου 2013, 4 και 5 Νοεμβρίου 2013, 28 Νοεμβρίου 2013, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις έως το τέλος της συνεδριάσεως, τα πρακτικά των ανωτέρων συνεδριάσεων λογίζονται εγκεκριμένα. Και προχωρώ στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα την έγκριση της απόφασης των συντονιστών που συνεδρίασαν σήμερα και συζητήσαν ε, την απόφαση της διασκέψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου για την πιθανή παρουσία του κυρίου Σνόντεν σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής μας για το θέμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καλούμεθα να υιοθετήσουμε την εξής απόφαση των συντονιστών. Να προσκληθεί ο κύριος Σνόντε να συμβάλλει στην έρευνα με μια ε, διαδραστική βιντεοδιάσκεψη και το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να προσκαλέσει τον κύριο Σνόντεν, ποιος είναι υπέρ, συγγνώμη, της πρόσκλησης για τον κύριο Σνόντεν να, έρθει, να συμμετάσχει με βίντεο διάσκεψη στις εργασίες μας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά παρακαλώ. Να επαληθεύσετε παρακαλώ. Καλώς ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρα στη σα. 36 υπέρ. 2 κατά. μια αποχή. Και άρα η απόφαση των συντονιστών εγκρίνεται από την Επιτροπή. Και προχωρώ στη ψηφοφορία τις προτάσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με συγγήτρια την κυρία Αντζελίλη και τη ρωτώ αν θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Απλώς να τονίσω ότι θα ψηφίσω αρνητικά για ορισμένα τμήματα των τροπολογιών 12 και 13. Θα ψηφίσω αρνητικά διότι κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να καταρτιστούν κατάλογοι όταν μιλούμε για θύματα. Δηλαδή κατάλογοι με τις κατηγορίες θυμάτων. Όλα τα θύματα βίων πράξεων είναι, πρέπει να την χάνουν ίσως μεταχειρήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν θύματα στα οποία θα αφοσιώνεται περισσότερη προσοχή. Όλες, όλοι οι κατάλογοι αποτελούν ε, αίτιο διακριτική μεταχείριση. Δεν μπορεί λοιπόν να προτιμάται μια κατηγορία ει βάρο μια άλλη. Θα πρέπει Λοιπόν, για αυτό το λόγο θα ψηφίσω αρνητικά. Now, let's to the vote. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Προχωρώ στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία τρίτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τέταρτη υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να υπολυθεύσω. Ψηφίζουμε την πρώτη παρακαλώ. Την τέταρτη τροπολογία. Πέρασε. 21 υπέρ, 22 κατά, αποχές δεν υπάρχουν, απορρίπτεται. Πέμπτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 σε τμήματα υπέρ, ε, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είκοσι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία Παρακαλώ κύριε Βερσία. Θα ήθελα πρόεδρε να ξανακοιτάξουμε κάτι γιατί από τον κατάλογο ψηφοφοριών δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέσατε σε ψηφοφορία τις τροπολογίες 12 και 13, οι οποίες όμως τα κατέπεπταν μόνο αν είχε υιοθετηθεί η 11, ενώ υιοθετήθηκε ανταυτής η συμβαστική 3. Στο δικό μου κατάλογο ψηφοφοριών, λέει ο πρόεδρος, λέει ότι καταπίπτει καταπίπτει 11 εάν υιοθετηθεί η 3. Και άρα αφού υιοθετηθεί η 3 δεν ψηφίσαμε την 11. Μα, κυρία Βεξιά, ε, ναι, αλλά η 12 και 13 μόνο αν ε, υιοθετηθεί η 11 δεν θα ψηφίζονταν με βάση τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Είσαστε εντάξει δηλαδή, λέει η πρόεδρος. Η γραμματεία μας λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 12. Τροπολογία 12. Σε δύο τμήματα. Άρα θα επανέλθω, αγαπητοί συνολφοί και στο συγγνώμη. Πρώτο τμήμα της 12, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε το πρώτο, μάλιστα. Πέρας. 27 υπέρ, 18 κατά, δύο αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν και ζητώ συγγνώμη. Το ίδιο ισχύει και για την 13 λέει η κυρία Βερζία. Τροπολογία 13. But Μα δε, η 13 καταπίπτει, λέει η πρόεδρος. τότε έχουμε πρόβλημα στο κατάλογο των ψηφοφοριών, γιατί δεν είναι σαφές. Πρέπει να ψηφίσουμε δηλαδή 13. Καλώς. Την ψηφίζουμε. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνομαι. Και σας ευχαριστώ. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά. Πέρας. 47 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή και συγχαρητήρια της στην κυρία Αντζελίλη. Και τώρα πάμε στην ψηφοφορία για επαλήθευση επιβεβαίωση των Γενικών Διατάξεων του Ταμείου για το Ασύλο και τη Μετανάστευση και του Ταμείου για την Εσωτερική Ασφάλεια. Έκθεση Φοντάνα καταρχάς. Uh, we vote on the compromise να ψηφίσουμε για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ξαναρωτήσω. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 40 υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάλι ψηφοφορία επιβεβαίωση για τα εξωτερικά σύνορα και τι θεωρήσει πάλι από το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια. Ο εισηγητή ο κ. Μαρινέσκου. Ψηφίζουμε το συμβαστικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία στο κείμενο που τροποποιήθηκε. Άρχεται. Πέρας. 36 υπέρ, 8 κατά, 4 εποχές. Αγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάλι ψήφος επιβεβαίωσης σχέδιο έκθεση για το Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια, Αστυνομική Συνεργασία, Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματο και Διαχείριση των Κρίσεων. Ο κ. Γιακολίνο, ηγητή. Θέλετε να σχολιάσετε. Ωραία. Ευθύ αμέσω ψηφίζουμε. Συμβαστικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο τον πήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παλήθευση. Πέρας. νέα πέρα, 8 κατά, 2 εποχές. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια, κύριε Γιακολίνο. Έχουμε άλλη μία. Άλλη μία. Ψήφο επιβεβαίωση, σχέδιο έκθεσης για το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, κυρία Κιγιόμ. Θέλετε να σχολιάσετε, Όχι. Ψηφίζουμε. Το συμβαστικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Πέρας. 45 υπέρ, 4 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια σου. Τελειώσαμε με τις προφορίες. Το επόμενο σημείο στην εμείς διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Φαγιών. Η οποία βέβαια ε, προβλεπόταν για τις 10.40. Θα πρέπει λοιπόν να διακόψουμε για λίγο μέχρι τις 10, μέχρι τις 11 παρά 20. Δεν είναι εδώ η συγκήτρια. Α, εκεί είστε. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Να συνεχίσουμε ή όχι μέχρι τις 10.40. Είναι εδώ η σκιώδη σας. <laughs> Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα ξαναρχίσουμε στις 10.40. Ευχαριστώ συναδελφοί. Τάνια, do you think we... Τάνια, πιστεύεις ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ωραία, λοιπόν. but, yeah, but I haven't seen Marinescu either for... Ο κ. Μαρινέσκου που είναι σκιώδης δεν ήταν εδώ ούτε στις ψηφοφορίες, οπότε δεν ξέρω. Να τον περιμένουμε, τι να πω. Ας συνεχίσουμε, ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το θέμα είναι οι τρίτε χώρε, οι οποίοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διάρκεια των εξωτερικών συνόρων και τρίτε χώρε οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Η συγκεκριμένη κυρία Φαγιών, για τη Μολδαβία μιλάμε τώρα, για την εξαίρεση ε, των υπηκών τη Μολδαβία, όταν ε, ταξιδεύουν εντό Σέγγεν, να κατέχουν ε, θεώρηση διαβατηρίου. Κυρία Φαγιών θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι συγγήτρια για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Διότι πιστεύω ότι στέλνουμε με τον τρόπο αυτό ένα πολύ χειρό μήνυμα στους πολίτες της Μολδαβίας. Η χώρα έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια μετά ε, το άνοιγμα του διαλόγου για την απελευθέρωση θεωρήσεων τον Ιούνιο του 2010 με τη Δημοκρατία του Μολδαβίας και είχαμε και ε, την έγκριση το ίδιο χρόνο του σχέδιου δράση για την απελευθέρωση θεωρήσεων. Στην περίοδο αυτή επισκέφθηκαν τη χώρα εμπειρογνώμονε, έκαναν μια αναλυτική, μια ανάλυση που επέτρεψε και την αξιολόγηση αυτού του διαλόγου για τις θεωρήσεις. Τρία χρόνια κράτησαν οι διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα ε, και με βάση τους στόχους του διαλόγου και των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων της χώρας εξέδωσε σύσταση για την υποχρέωση ε, θεώρησης ε, η οποία έρεται για τη δημοκρατία της Μολδαβίας εφόσον όλα τα κριτήρια πληρούνται. Επίσης έχουν διατεθεί και οι επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, ώστε να είναι βιώσιμες οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Σήμερα χαίρομαι που βλέπω ότι η Μολδαβία είναι η πρώτη χώρα της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που κάνει τα πρώτα πολύ σημαντικά της βήματα προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Ο διάλογος για τις σα ε, τα τελευταία χρόνια ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μολδαβία. Θα ήθελα επίσης να ε, τονίσω ότι για, την, ε, για τους ανθρώπους τους απλούς είναι το πιο μεγάλο όφελος. Πολλά είναι τα ωφέλη για όλους τους απλούς πολίτες με την απελευθέρωση της θεώρησης, θα μειωθούν ε, οι χρόνια αναμονής στα γκισέ, το κόστος ε, ταξιδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διευκολυνθούν διαπροσωπικές επαφές, που είναι και σημαντική προϋπόθεση για μια σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ε, επιστημονικών και άλλων δεσμών. Ελευθερία κυκλοφορία επίση διευκολύνεται και ξέρουμε ότι αυτή είναι μια από τι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία τη εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ τη Ένωση και τη Μολδαβία αναμφίβολα θα συνεισφέρει στη βελτίωση ε, τη άσκηση ε, ε τη δικαιοσύνη και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. όπω είπα και στην αρχή είναι σημαντικό να εκπέμψουμε ένα ηχηρό και πολύ ε, ξεκάθαρο μήνυμα προς τους κατοίκου της Μολδαβία, ιδιω τώρα με την πρόσφατη εξέλιξη που είχαμε στην ε, περιοχή την ευρύτερη και λόγω βέβαια της πολιτικής και γεωστρατηγικής κατάστασης της χώρας, η Μολδαβία έχει καταδείξει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η μόνη εναλλακτική για τη χώρα. Και ελπίζω ότι με το βήμα αυτό η Μολδαβία θα συνεχίσει το ταξίδι της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εισηγητρία ε, καλωσορίζω θερμά την πρόταση της ε, Κομισιόν και δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη για κατάθεση περαιτέρω τροπολογιών. Ο στόχος μας είναι μια ομαλή γρήγορη έγκριση τη έκθεση στο Κοινοβούλιο και φαντάζομαι ότι θα γίνουν ε, όλα τα πάρτα βήματα και θα ληφθούν τα πάρτα μέτρα και σε επίπεδο Συμβουλίου ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα πριν τις ευρωεκλογέ του Μάιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σκουέλιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λυπάται ο κύριος Μανέσκου που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, πάντως μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο μετά τη Βενετία πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία της ε, αυτοεξωτερικής σχέσης ε, και πόσο σημαντική είναι αυτή, παραδείγματος για τη δημοκρατία της Μολδαβίας, η οποία έχει ε, περάσει με τεχνική μεταρρύθμιση για την εκπλήρωση κάποιων κριτηρίων, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση της, των θεωρήσεων μετά τη 15η, 11η και τις αξιολογήσεις που έγιναν βλέπουμε ότι υπάρχουν απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Στο σχέδιο δράσης ε, ε, είχαν ε, περιληφθεί μεταρρυθμίσεις, έγιναν δράσεις εκτίμησης αξιολόγησης και βλέπουμε ότι πληρούνται πολλοί οι όροι και έχουν ξεπεραστεί και προηγούμενες τέτοιες διαδικασίες όπως αυτή Δυτικά Βαλκάνια. είναι φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας. Βλέπουμε ότι έχει εκπληρώσει τα κριτήρια των τεσσάρων ε, δεσμών της πρώτης και δεύτερης φάσης ε, του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των ορίσεων. Η Μολδαβία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ε, για να εκπληρώσει όλους τους όρους και προϋποθέσεις με την αποτελεσματική σταθερή εφαρμογή Παρακολουθεί καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές, δημιουργεί, έχει δημιουργήσει περιφερειακά γραφεία για τη μετανάστευση. Επίσης έχει κάνει προσπάθειες για τη σύναψη επιχειρησιακών συμφωνιών με τη Europol και τη Eurojust. Και υπάρχουν και τα πρότυπα ασφαλείας τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκδοση διαβατηρίων είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ECO και είναι κάτι το οποίο δεν τήρουν άλλες χώρες περιοχής έχουν δημιουργηθεί κινητέ μονάδες για την επίβλεψη των ε, επιτυγμένων εδαφών εντό και εκτός επικράτειας. Σε ό,τι αφορά τώρα τι επιπτώσει που θα έχει η απελευθέρωση θεωρήσεων, στον τομέα τη μετανάστευση και τη ασφάλειας έκανε η Κομισιόν μια σχετική ε, εκτίμηση. Υπάρχουν, υπάρχει συνεργασία στον τομέα τη μετανάστευση Υπάρχει συμφωνία για την διευκόλυνση θεωρήσεων και γενικά όλα αυτά έχουν διευκολύνει πολύ την κατάσταση. είναι ικανοποιητική εκτέλεση της συμφωνίας ε, για τη διευκόλυνση θεωρήσεων από τη Δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Ο διάλογος επίσης ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Και ο κ. Βανέσκο θεωρεί εν κατακλείδη ότι η πρόοδος της Μολδαβίας στην τελευταία τριετία αποδεικνύεται με τις μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς. Έχουν μειωθεί οι αρνήσεις ε, χορήγησης θεωρήσεων και λόγω της εργασίας, όπως είπα στο προηγούμενο μου σημείο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες ε, του Κισινάου και βέβαια να εξασφαλίσει ε, ότι θα παραμείνει ε, στο δρόμο τον Ευρωπαϊκό η Μολδαβία. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος, η κυρία Ντανόκα. Thank you. Ευχαριστώ. Να πω καταρχάς ότι η ομάδα μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων ιδίως ό,τι αφορά τους ανατολικούς γειτονές μας και εταίρους. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Όταν απελευθερώνεται το καθεστώς θεωρήσεων, πολλές φορές υποκρύπτονται και πολιτικοί πολιτικές σκοπιμότητες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να το συζητήσουμε όπως έχουμε κάνει στην πολιτική μας ομάδα. Μήπως δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική θεωρήσεων για ακριβώς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ίσως να ήταν προτιμότερο να υπάρξει απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων ταυτόχρονα με όλες τις ανατολικές χώρες και τη Ρωσία. Μόλις ε, ήρθα από μια συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και την ε, συνεδρίαση προφανώς της αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας όπου συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Μολδοβία. Ξέρω πολύ καλά την κατάσταση στη χώρα αυτή. Και ξέρω ότι οι περισσότεροι Μολδαβοί οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ρουμανικά διαβατήρια. Κάποιες φορές έχουμε περισσότερο ε, κατόχους μολδαβικών διαβατηριών στους κατοίκους της υπερδυναστερίας. Άλλωστε, οι περισσότεροι Μολδαβοί υπήκοοι έχουν διπλή υπηκότητα, είτε και ρουμανική και ουκρανική ή και ρωσική. Η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη λοιπόν. Και δεν λέω να μην διευκολύνουμε, να μην απλοποιήσουμε και απελευθερώσουμε το καθεστώ θεωρήσεων το, για του Μολδαβού πολίτε, ακόμη και αν είναι κάτω ρουμανικών διαβατηρίων. Όμω πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε μια εναρμονισμένη πολιτική για τα θέματα αυτά. Βεβαίω η συζήτηση έχει πολιτικέ ε, διαστάσει. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συζητηθεί και στι στις πολιτικές ομάδες και γενικώ στο Κοινοβούλιο. Είναι πάντω ένα ζήτημα περίπλοκο. Και κύριε Κοέλιο, θα ήθελα αντί να τα λέω σε εσά, να τα πω στον ίδιο τον κύριο Μαρινέσκου. Δεν ξέρω αν εσεί μπορείτε να απαντήσετε στη θέση του κιόλα, αλλά υπήρξαν κάποια σχόλια στην παρέμβασή σας Και ξέρουμε ότι θα διοργανωθεί τριμερής διάλογος σύντομα για το θέμα αυτό και θα διοργανωθεί, θα, θα υπάρξει έγκριση του σε αυτό. Λοιπόν, δεν συμφωνώ για τα σχόλια, με τα σχόλια του κ. Μαρινέσκου για τους Μολδαβούς πολίτες, όμως θα πρέπει να συζητήσουμε το όλο θέμα σε επίπεδο ομάδας, διότι τα περισσότερα σχόλια μου τώρα σήμερα ήταν πολιτικά, προσωπικά, αλλά θα φροντίσω να εκφράσω και την άποψη της ομάδας μου. Ευχαριστούμε κυρία Ντανόκα. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Ένα λεπτάκι. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά μια και μίλησα για εναρμονισμένη πολιτική περιθεωρήσεων, να μην ξεχνάμε τα Βαλκάνια και το πρόβλημα του κοσφοπεδίου. Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία της παρουσίας της Επιτροπής εδώ να θυμίσω ότι οι πολίτε του κοσμοπεδίου δεν ε, έχουν τη δυνατότητα ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν υπήρχε ένα κοινό διάγραμμα για όλε αυτέ τι χώρε τη Ανατολική Συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στρέφομαι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστώ με ειλικρίνεια την εισηγήτρια για την πλήρη υποστήριξη που προσφέρει στην πρόταση Επιτροπής. Και όντως πιστεύω ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατευτεί για τον διάλογο αυτόν, για την απελευθέρωση από την υποχρέωση των δημοτηρίων με τι γειτονικές χώρε, θα πρέπει και να τιμήσει τις ε, δεσμεύσεις της. Η Μολδοβία έχει κάνει ό,τι όφιλε, πλήρει όλους τους όρους για την απελευθέρωση και γι' αυτό αμέσως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει την πρόταση εκείνη η οποία εκπληρώνει το μερίδιο της ε, συναλλαγής της ε, συμφωνίας εκ μέρους ευρωπαϊκής πλευράς. Και χαίρομαι που και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασφαλώς θα μιλήσει σε λίγο. Ε, συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση και ανταποκρίνεται στις ε, προσδοκίες αυτής της χώρας. Και αν το ολοκληρώσουμε από πλευράς μας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση. Και για να απαντήσω στη τελευταία παρέμβαση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο διάλογος για την απελευθέρωση είναι διάλογος ο οποίος στηρίζεται στην αξιολόγηση των συνθήκων σε κάθε χώρα χωριστά. Έτσι έγινε και με τη Μολδαβία. Μελετήσαμε με βάση τα τέσσερα ε, πακέτα, τα τέσσερα κεφάλαια που προβλέπονται για την απελευθέρωση και διαπιστώσαμε ότι για τη Μολδαβία συντρέχουν οι όροι άρση τη υποχρέωση. Το ίδιο θα γίνει αργότερα και για το κοσμοπέδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν χορηγείται η απελευθέρωση, η άρση τη υποχρέωση για μια χώρα πρέπει να αναγνωρίζεται και για τι υπόλοιπε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προ το παρόν, επειδή αξιολογούνται πάντα χωριστά η κάθε μια χώρα, έχει έρθει η ώρα για την Μολδαβία να υποβληθεί η σχετική τρόπαση, πρόταση αφού αυτή πληρεί τις υποχρεώσεις και έτσι θέλουμε να άρουμε την υποχρεώση για θεώρηση ώστε και οι πολίτες της Μολδαβίας να επωφεληθούν αυτής της ευχέρειας ταξιδιών. Επί της ουσίας ένα πράγμα θα ήθελα να φέρω ότι στο Συμβούλιο ξέρουμε ότι εν γέννη επικρατεί υποστήριξη για την πρόταση. Υπάρχουν όμως κάποια κρατημέλη τα οποία εκφράζουν σε σχέση με τα βιομετρικά διαβατήρια που αναπτύσσουν τώρα οι αρχές της Μολδαβίας ε, κάποιες επιφυλάξεις. Γιατί? Γιατί είναι διαβατήρια τρίτης γενιάς και άρα μέσω ενός στίκερ, ενός αυτοκόλλητου δηλαδή μπαίνουν ε, πάνω στο διαβατήριο. Δεν είναι δηλαδή της τελευταίας ε, τεχνολογίας τα διαβατήρια που προβλέπονται προς το παρόν. Ωστόσο η Μολδαβία μας λέει ότι είναι έτοιμη να εκδώσει διαβατήρια τετάρτης γενιάς όπου το μικροτσίπ είναι ενσωματωμένο στο ε, εξώφυλλο του διαβατηρίου και άρα προσφέρει αυξημένη ασφάλεια. Αλλά κράτη μας λένε ότι μπορούν ε, να... Ε, η Μολδαβία μας λέει ότι είναι σε θέση να αρχίσει αμέσως να εκδίδει αυτά τα βιομετρικά διαβατήρια τέταρτης γενεάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πληρεί τις υποχρεώσεις της για την άρση των ε, τις υποχρεώσεις θεώρησης. Απλώς για να απαντήσουμε εμείς στις επιφυλάξεις κάποιων κρατών, είμαστε διατεθειμένοι ως Επιτροπή, κατά τη στιγμή της υιοθέτησης προτάσεως, να εκδώσουμε την εξή ανακοίνωση. Και παραθέτω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει την κυβέρνηση της Μολδαβίας την απόφαση την οποία έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση της Μολδαβίας για την εισαγωγή των ε, για την αντικατάσταση καλύτερα των διαβατηρίων Τρίτη γενεάς που προβλέπονται για του πολίτες τη από διαβατήρια τετάρτη γενεάς βιομετρικά, η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί 2000, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή του το 2015 και ε, εξακολουθεί να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πλαίσιο και την υλοποίηση των ε, αποφάσεων με βάση το διαρθρωμένο διάλογο και θα εξακολουθήσει να αναφέρεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την υλοποίηση της απόφαση αυτή στο πλαίσιο τη εκθέσεω παρακολούθηση Τη τη υλοποίηση απόφασης περί ε, Αυτό λοιπόν ω μια ανακοίνωση μόνο ότι θα παρακολουθούμε τι προσπάθειες των αρχών τη Μολδαβία και την πορεία του στην ε, ε, έκδοση των βιομετρικών διαβατηρίων τετάρτης γενιά. Και τώρα ερωτώ, λέει η πρόεδρο την ελληνική Προεδρία αν θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με χαρά ενημερώνω την Επιτροπή σας ότι χάρη και στην Λιθουανική Προεδρία μπορέσαμε να έχουμε μια επικοδομητική προσέγγιση στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου, για την μεταφορά της ε, χώρας της Μολδαβίας στον θετικό κατάλογο. Αυτό χωρίς αλλαγές οι δε επιφυλάξεις που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη ως προς την ασφάλεια των βιομετρικών διαβατηρίων που εκδίδει η Δημοκρατία της Μολδαβίας αντιμετωπίστηκαν με τον τρόπο που σας εξήγησε μόλι τώρα εκπρόσωπος Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, ο κάθε ένας από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει τη μεγάλη σημασία της ε, ταχείας διεκπαιρέωσης του φακέλου αυτού ώστε να έχουν οι πολίτες της Μολδαβίας ένα καθεστώς χωρίς θεώρηση διαβατηρίων το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε διατεθειμένοι σε ελληνική προεδρία να συνεργαστούμε όσο δυνατόν πιο εντατικά με την κυρία Φαγιών αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρωθεί το ζήτημα αυτό το ταχύτερο δυνατό και να προσφέρουμε στου πολίτε τη Μοσλαβία την ευχέρεια της ε, διακίνηση των ταξιδιών χωρί την υποχρέωση θεώρηση. Ευχαριστώ κύριε και έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Γιατί στις 11 πρέπει να είμαστε σε άλλη αίθουσα πολύ σύντομα. Για το κοσφοπέδιο, το, το ερώτημα των συναδέλφων, επειδή είμαι και εισηγήτρια στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Το θέμα δεν είναι να μην ε, είναι βασισμένο ε, στην αξία, το, λεγόμενο merit-based. Και οι προσπάθειες του κοσφοπεδίου πρέπει να ε, κάνουν περισσότερες προσπάθειες, θα το δείτε και στο Στρασβούργο στην εκθεσή μου, τα λέω. Το θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα με τις επισκέψεις του κοσφοπέδιου ήταν ε, πολύ ε, πιο φορτωμένο το πρόγραμμα και κρατά πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή νιώθουν οι πολίτες του Κοσμοπεδίου ότι έχουν διαφορετική μεταχείριση, παρότι παραδίδουν αποτελέσματα, προχωρούν. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό ήθελα να απαντηθεί από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ε, κυρία Λότσε και κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για μια κομφρά να πω ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι κάτι απτό για τους πολίτες, άρα είναι άκρος ε, λεπτό πολιτικό ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να είχαμε περισσότερη ώρα στη θέση να το συζητήσουμε, γιατί σήμερα άνοιξαν πολλά θέματα ε, που αφορούσαν μεταξύ άλλων και το Κοσμοπέδιο και Βαλκάνια. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα, ο νέος μηχανισμός για την προσωρινή αναστολή ε, του καθεστώτο θεωρήσεων τίθεται σε ισχύ και αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ειδικά σήμερα νιώθουν ότι θα είναι οι πρώτες που ίσως ε, ξαναπάρουν ή ξαναέχουν αυτή τη που χρειάζεται τις θεωρήσεις ε, τις επόμενες μέρες και μήνες και υπάρχει μεγάλη πίεση, δημαγωγία, λαϊκίστικη ε, πίεση για κατά τον μεταναστών και τον άσυλο. Συμφωνώ βέβαια με τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε και να ζητούμε όλες οι χώρες που ζητούν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώ, ε, το απαλλαγμένο από δηλαδή, για όλες τις χώρες να ισχύουν τα ίδια κριτήρια. Επίσης, χθε ακούσαμε ε, ότι σε ένα τριμερή διάλογο που συζητούσε ε, το Περού, την Κολομβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κάποιες άλλες χώρες. δεν θέλω να μπω σε άλλη τώρα συζήτηση, αλλά Νομίζω ότι αξίζει η Μολδαβία να μπει ε, στο καθεστώς ε, ως επόμενη χώρα. Γιατί μέσα σε μια τριετία έχουν κάνει πάρα πολλά για να εκπληρώσουν όλα τα κριτήρια. Αυτή η διαδικασία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη είναι μια διαδικασία που πρέπει να ισχύσει και για τους υπόλοιπους στο μέλλον. Η Κομισιόν πρέπει να έχει και μια συνεπή στάση. Και το ίδιο που έκανε με τις προηγούμενες χώρες να τα κάνει και με το κοσυφοπαίδιο. Συμφωνώ και εγώ ότι είναι πολύ πιο χρονοβόρα η διαδικασία που ακολουθεί για το κοσυφοπαίδιο και θεωρώ επίση ότι είναι πολύ σημαντικό εμεί, στην Επιτροπή μα ιδίω, αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικά να επιχειρηματολογήσουμε με όλη μα τη δύναμη ε, για το πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτική απελευθέρωση θεωρήσεων και για τις ε, γείτονε χώρε, διότι ενισχύει όχι μόνο την πολιτική και οικονομική συνεργασία, αλλά και τις διαπροσωπικές επαφές των πολιτών πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαγιόνλη Πρόεδρος. Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ε, επί του σημείου αυτής της μερικής διάταξης και θα ζητήσω από τους αδέλφους να έρθουν σε μια κοινή συνεδρίαση ε, με την Επιτροπή Οικονομικών στην αίθουσα 4Q1 για την ε, πρόληψη της κρίσης του ψηφιακού συστήματος για σκοπούς ξεπλήματος χρήματος. Έχουμε προθεσμία για την έκθεση φαγιών για την κατάσταση τροπολογιών που τώρα ορίστηκε 30 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Συνάδελφοι, ευχαριστώ και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στην ε, αίθουσα 4Q1.